Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, Πάτης εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας με θέμα Γουινέα Μπισάου. Εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και της ε, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας το λόγο έχει ο κύριος Νικολάη Βάμεν. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι ευτυχή για την ευθερία να συζητήσω σήμερα μαζί σας εξ ονόματος της ΥΠΕΤ προσώπου της Αντιπρόεδρου Αύστον την κατάσταση στη Γουινέα Μπισάου και χαιρετίζω την προσοχή που δίνει στο θέμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τρέχουσα κρίση στη Γουινέα Μπισάου αποκαλύπτει ακόμα μια φορά σαφώ μια προσπάθεια του ερωτικού να εμπλακούν στι υποθέσει των πολιτών και να αποκτήσουν τον έλεγχο των πολιτικών υποθέσεων στη χώρα. Η χώρα παραμένει μια φτωχότερο στον κόσμο, μαστίζεται από λαθρεμπόροι ναρκωτικών και τα προβλήματά τη άμεσα επηρεάζουν την Ευρώπη μέσω αυτού του λαθρεμπορίου η λύση είναι να πιστούν οι στρατιωτικοί να αποχωρήσουν και να προβούν σε μεταρρυθμίσεις του στρατού. Μόνο τότε η χώρα θα μπορεί να κυβερνείται από, κυβερνάται από πολίτες που θα έχουν νομιμοποιηθεί μετά από ελεύθερες και αδιάβλητε εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την πραξικόπημα στη Γουινέμπισα τη της 12 Απριλίου 2012 και ζητά την άμεση επιστροφή της νόμιμης κυβέρνησης και την διεξαγωγή προεδρικών εκλογών σύμφωνα με την νομοθεσία. Χαιρετίζουμε την ομόφωνη ψήφιση στις 18 Μαΐου του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματος 2048-2012 για τη Γουινέα Μπισάου και τις επιβολής που επιβάλλει ατομικές κυρώσεις για τους υπεύθυνους, στους υπεύθυνους του πραξικόπηματος και αποτά, απαιτεί την άμεση αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης συμπεριλαμβανομένης και μιας δημοκρατικής εκλογικής διαδικασίας, την επιστροφή των στρατιωτικών στις βάσεις τους και την απόσυρσή τους, απομάκρυνσή του από τις πολιτικές υποθέσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογράμμισε ότι εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν και ότι μία μόνιμη λύση για την αστάθεια στη Γουνέα Μπισάου θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ε, όσοι ήταν υπεύθυνοι για τι δολοφονίε για πολιτικού λόγου και άλλα σοβαρά εγκλήματα και παραβιάσεις τη συναματική τάξη να προσταχθούν στη δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνουμε την ισχυρή καταδίκη μα ε, για το πραξικόπημα και καλούμε όλου του ενδιαφερόμενε πλευρέ να συνεργαστούν μέσα στο πλαίσιο και σύμφωνα με το ψήφισμα 28 2048 των Ηνωμένων Εθνών ώστε να συμφωνήσουν για, μια, για έναν χάρτη πορείας με σταθμούς συμφωνημένους και ένα χρονοδιάγραμμα έως ότου αποκατασταθεί συνταγματική τάξη στη χώρα την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας, την καταπολέμηση της ατιμορρησίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και την απομάκρυνση της, ε, εξουσία, της ισχύς των στρατιωτικών στη χώρα. Επαναλαμβάνουμε την ε, έτοιμά μας για άμεση απελευθέρωση όλων εκείνων που κρατούνται παράνομα συμπεριλαμβανομένων και των μελών της πρώην Και ζητούμε από τα μέλη της πρώην κυβέρνησης να αναχωρήσουν από τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ε, εφαρμόσει κυρώσεις παγώνοντας ε, τις καταθέσεις και απαγορεύοντας τα ταξίδια εναντίον έξι μελών της στρατιωτικής διοίκησης και είναι τετεθειμένη να επεκτείνει τον κατάλογο αυτό σε άλλα άτομα, στρατιωτικούς και πολιτικούς που κυβερνούν τη χώρα de facto και μπορεί να είναι υπεύθυνοι για παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά χρήσεων παντός τύπου αυθαίρετων κρατήσεων κλπ. Μας ε, απασχολεί επίσης η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση και ο κίνδυνος βίας. Μας απασχολεί επίσης η δυνατότητα διευθετήσεων που θα επιτρέπουν στους σημερινούς ηγέτες του στρατού να εξακολουθούν να απειλούν ή να ελέγχουν τις πολίτες. Η δημοκρατική σταθερότητα στη Γουινέα Μπισάου απαιτεί την απομάκρυνση της απειλής που εκπροσωπούν οι ένοπλες δυνάμεις και η μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλεία παραμένει επίγουσα ανάγκη. Όσοι είναι υπεύθυνοι για την αντισυνταγματική συμπεριφορά ή για εγκλήματα πρέπει να λογοδοτήσουν. Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει όλου και να είναι δημοκρατική. Οι στρατιωτικοί δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπαγορεύουν ποιο θα συμμετέχει και ποιο δεν θα συμμετέχει στα πολιτική ζωή του τόπου. Παρακολουθούμε τι πρόσφατε πολιτικέ και ε, ε, ε, εξελίξει και τα θέματα ασφάλεια υπό αυτό το πρίσμα. Η διεθνή διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει ενωμένη. Από την άποψη αυτή, η ΑΕΠΑΤΗ εκπρόσωπος κάλεσε την ECOWAS και την Αφρικα... Ε, Αφρικανική Ένωση να συναντηθούν ε, να ε, συγκαλέσουν όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές της διεθνούς κοινότητας σε μία συνάντηση ώστε να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες για την εφαρμογή του χάρτη πορείας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, πρώτος στον κατάλογο, εξ ονόματος της κοινωνιστικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Δημοκρατών, ο συνάδελφος κύριος Πάουλο Ρανζέλ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, Βάνεν. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι αξιοθρύνητο που σε μια τόσο σημαντική συζήτηση απουσιάζει η ύπατη ε, και την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Άστον. Πάντω, έχουμε την ευκαιρία να συνεργαζόμαστε για μια ακόμη φορά με τον Υπουργό Βάνεν ε, που έκανε τη δήλωση που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ε, υποστήριξη και την αλληλεγγύη μου προς το λαό της Γουινέας, ένα λαό που έχει ε, δυνοπαθήσει από την δημοκρατική αστάθεια, από την πολιτική αστάθεια και την ανασφάλεια που επικρατεί. Δεν είναι μόνο η φτώχεια και η εξαθλίωση, ε, από πολλά δεινά έχει πληγεί ο λαός της Γουινέας και μάλιστα το ΕΛΚΑ ε, από την αρχή παρακολούθησε αυτό το θέμα και είναι κρίμα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο μετά από ένα μήνα σε ε, να οργανώσει συζήτηση για το θέμα αυτό. Βλέπετε πόσο, ποια, τι άγνοια υπάρχει για το λαό της Γουινέας Μπισάου και για την ίδια τη χώρα ε, τη Γουινέα Μπισάου. Γιατί εδώ δεν έχουμε σημαντικά οικονομικά συμφέροντα, δεν έχουμε κίνητρο ε, των κυβερνώντων και των σημαντικών χωρών για να ασχοληθεί με τη Γουινέα Μπισάου. Γι' αυτό και είναι αόρατη, ανύπαρκτη από τη διεθνή ατζέντα. Ε, χρειάζεται να έχουμε εξαθλίωση και πολιτική αστάθεια για να αναλάβουμε κάποια δράση. Έχουμε τέτοια, ε, τέτοιο λαθρεμπόριο ναρκωτικών που ξεκινάει από την Γουινέα Μπισάο ε, και ε, πλήττει τελικά τους, τον Αμερικανικό λαό και τους Ευρωπαϊκούς λαούς. Χρειάζεται να επικαλεστούμε αυτό το επιχείρημα για να αναλάβω μια δράση για τη Γουινέα Μπισάο. Είναι αναφυσβήτητο ότι οι αποφάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ε, Αφρικανικής Ένωσης, της ΕΚΟΒΑΣ ε, είναι σημαντικές και βρίθουν αγαθών προθέσεων, αλλά δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε ευχολόγια. Θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με στενή συνεργασία με τις χώρες που έχουν δυνατότητα παρέμβαση στη Γουινέμπισα. Αυτή είναι δική μας υποχρέωση και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, είναι εντάξει στη, σε επίπεδο αρχών και ε, διακηρύξεων, αλλά δυστυχώς υστερεί η δράση της σε πρακτική, στην, στην καθημερινότητα. γλώσσα ε, συνέχεια, πορτογαλικής παρουσίας συνέχεια, εξ της ομάδας Προδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Άννα Γκόμες για δύο λεπτά. Για δυόμιση λεπτά, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου για το λαό της Γουινέας που έδωσε τόσα μαθήματα στον κόσμο και σε μένα προσωπικά σε ό,τι αφορά τη, τον αγώνα κατά της απικιακής, απικρατικής καταστολής. Δυστυχώς ε, κάναμε ένα λάθος ε, με την απόσυρση της ενίσχυσης και απόσυρση της βοήθειας στο τομέα ασφάλειας ε, μετά από τις πολιτικές δολοφονίες του 2010. Ήταν τότε η στιγμή που έπρεπε να ενισχύσουμε την εντολή της αποστολής αντί να την αποσύρουμε. Όπως είπε ο Υπουργός Βάνεν, αυτό που ε, χρειαζόταν είναι να γυρίσουν οι στρατιωτικοί στους στρατώνες και να αναλάβει την εξουσία ο πολιτικός κόσμος. Χρειαζόμαστε συνταγματική τάξη και ασφάλεια για τους πολίτες. Δεν πρόκειται ο στρατός να ενισχύσει την πολιτική διακυβέρνηση γιατί ουσιαστικά θα εξυπηρετήσει το οργανωμένο έγκλημα και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτικά και στην πράξη και όχι μόνο στη, στα χαρτιά το ψήφισμα 2048 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εκεί κατονομάζονται οι πραξικοπηματίες, επιβάλλονται κυρώσεις και ζητείται επαναφορά της εξουσίας ε, στον Πρωθυπουργό του Ζούνιορ και τον, τον μεταβατικό πρόεδρο Περέιρα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις φυλακές. Επίσης θα πρέπει ε, να ζητήσουμε στην ΑΚΕ να αναλυθεί κάποια δράση γιατί έχουμε διατρανώσει την προσήλωσή μας προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν ε, η CDO να, ε, να δέχεται λύσεις που ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι των πραξικοβιομετειών, καταστρατηγώντας τη συνταγματική τάξη. Η Γουινέα Μπισάου είναι επίσης εταίρος στην ΑΚΕ. Δεν μπορεί να μένει εγκαταλειμμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με, το με τον ΟΗΕ, με την Αφρική, Αφρικανική Ένωση και με τη CPAP για να διασωθεί αυτή η χώρα που βρίσκεται στο χείλος της αναρχίας με εξαθλίωση, με έλλειψη διακυβέρνησης και κατασπατάληση των φυσικών πόρων. Η... Θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την ανάκτηση της εξουσίας από τον Πρωθυπουργό, έστω και στρατιωτικά. Χρειαζόμαστε μια συντονισμένη πολιτική και να προστατεύσουμε το λαό της Γουινέας Μπισέου από μια επικείμενη ανθρωπιστική τραγωδία και επίσης να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα δράσης για να εκριζωθούν τα αίτια του κακού που είναι η πανάπτυξη, η εξαθλίωση και η έλλειψη διακυβέρνησης. Θα πρέπει να δώσουμε το παρόν γιατί η ασφάλεια της Γουινέας Μπισάου σχετίζεται και με τη δική μας ασφάλεια, ε, με τη δρομοκρατία και με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ευχαριστώ εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας ο συνάδελφος κύριος Ρουί Τάβαρες. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από ένα μήνα είπε ότι εκπρόσωπο η κυρία Άστον ήταν εδώ στη συζήτηση και της εξέφρασα την ε, θλίψη μου γιατί ενώ για τη Ρεψόλ ε, ήταν άμεση η αντίδρασή της για τη Γουινέα Μπισά δεν ε, είπε τίποτα. Ε, τι περιμένουμε για να λάβουμε δράση για την Γουινέα Μπισάου. Βλέπουμε ότι ένα μήνα μετά ε, δεν είσαι καν να παρίσταται στη συζήτηση, είπατε εκπρόσωπο. Είναι πραγματικά αξιολείπητη η κατάσταση αυτή. Επιβεβαιώνω αυτή, αυτό που είπε ο κ. Ραζέλ. Είναι αόρατη η Γουινέα Μπισάου από το παγκόσμιο προσκήνιο. Υπάρχει έλλειψη ευαισθησία για τα προβλήματα τη χώρα αυτή. Ο λαό τη Γουινέα Μπισάου κάνει ό,τι μπορεί για να αποφευχθεί να γίνει άναρχο το κράτο τη Γουινέα Μπισάου. Δυστυχώ, οι στρατιωτικοί συνεργάζονται με τους λαθρεμπόρους ναρκωτικών και θέλουν ένα τέτοιο άναρχο κράτο. Χρειαζόμαστε επέμβαση τη παγκόσμια κοινότητα για να λυθούν τα προβλήματα. Ε, μάλιστα, ο Πρωθυπουργό ε, τη ε, Γουινέα Μπισάου έχει πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Πορτογαλία για να ζητηθεί βοήθεια να αποφευθεί η ανάληψη τη εξουσία από του πραξικοπηματίε. Είναι σωστό το ψήφισμα 2048 του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ και συμφωνώ με αυτά που είπε ο εκπρόσωπο τη ε, εκπροσώπου. Το θέμα δεν βρίσκεται σε επίπεδο ευχολογίων και ρητορική, αλλά σε επίπεδο πράξεων. Θέλουμε ε, συνάντηση υψηλού επίπεδου με, τους, ε, με την ΕΚΟΒΑΣ, την Οικονομική Κοινότητα Χωρών της Δυτικής Αφρικής. Θέλουμε αποδοχή της ε, πρότασης για διορισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης και εφαρμογή του ψηφίσματος ασφαλείας στο ΙΕ. Να αποσταλεί βοήθεια δύναμη σταθεροποίησης και ειρήνης, να υποστηριχθεί η ανάληψη εξουσίας από την νόμιμη κυβέρνηση και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάποια λάθη που κάναμε όπως ήταν η απόσυρση της κοινοτικής αποστολής του Γουινέα Μπισά προκειμένου να βοηθήσουμε ε, την μετάβαση ή ε, την την, ε, τον εξυγχρονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων, την ε, πιο πολιτιστική, πολιτιστική τους δράση, προκειμένου να, η, να επανέλθει η Γουινέα στο σωστό δρόμο. Ευχαριστώ. ...της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο συνάδελφος κύριος Τσάρλς Στάνοκ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, από τότε που απέκτησε την δεκαετία του 70 την ανεξαρτησία από την Πορτογαλία, αυτή η φτωχή χώρα ε, στη Δυτική Αφρική βρίσκεται σε ένα καθεστώ σχεδόν μόνιμη σύγκρουση ενό εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στου πολίτε ε, και την στρατιωτική εξουσία. Η δική μου ομάδα ε, καταδικάζει τα τελευταία γεγονότα τον τελευταίο μήνα, όπου ανετράπη η κυβέρνηση και επικράτησε η Χούντα. Ε, πρέπει λοιπόν ε, να ε, επενέσουμε την προηγούμενη κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας και να ε, υπάρξουν ουσιαστικές ε, διαπραγματεύσεις, απειλές ε, οικονομικών κυρώσεων. Αυτά κατόρθωσαν επιτέλους να σπάσουν το αντιέξοδο και να σταθεροποιηθεί η χώρα. Άκουσα ότι παρετείται σιγά σιγά η Χούντα και παραδίδει σε πολιτική κυβέρνηση με ελπίζω την, το ενδεχόμενο ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ζητήσει από την υπηρεσιακή κυβέρνηση να προβεί σε μεταρρυθμίσει να ξεχνάμε ότι μια δημοκρατική γουένα είναι προς όφελος της Δύσης. Η χώρα δυστυχώς ε, είναι ο κόμβος ε, για μεταφορά νεροκατοικών από την Κολομβία προς την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν ο αγώνας ε, κατά των ε, παράνομων ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος ε, συνεχίζεται. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση και να ασκήσει κυρίως οικονομική πίεση προς την Γουινέα Μπισάου για να αντιδράσει αυτή λογικά να είναι ένα κράτος φυσιολογικό και όχι ένα αποκαλούμενο κράτος ναρκωτικών. τα Ηνωμένα Έθνη με τη δική μας τη βοήθεια πρέπει να προχωρήσουν έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα για όλου του πολίτε. Σύμφωνα με τον κύριο Ταβάρε ότι αν δεν μπορεί να είναι εδώ η κυρία Άστον, δυστυχώ βέβαια, γιατί ο κύριο Westcott που είναι διευθυντή για την Αφρική δεν ήρθε εδώ για να παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση. Τάνοκ, ολοκληρώθηκε ο κατάλογο των ομιλητών εξ ονόματο των ε, πολιτικών ομάδων και ανοίγει αυτός των άλλων εγγεγραμμένων ομιλητών. Πρώτος είναι, ε, στον κατάλογο είναι ο κύριος Διόγκο Φέιο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η συζήτηση που κάνουμε σήμερα βασίζεται σε ένα συμβάν της 12 Απριλίου τότε που ο στρατός ανέλαβε καταχρηστικά την εξουσία με ένα ε, πραξικόπημα και φυλάκισε ε, τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό και ε, ανέθεσε την εξουσία σε ένα εθνικό συμβουλίο χωρίς καμία δημοκρατική και πολιτική νομιμοποίηση. Ε, το κράτος της Γουινέας Μπισάου βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Πρόκειται για ένα έθραυστο κράτος, ένα κράτος που χρήζει υποστήριξης και αρρωγής για να περάσει σε μια κατάσταση νομιμότητας και νομιμοποίησης. Γίνονται πολλές διαμαρτυρίες από τη διεθνή κοινότητα. Οι περισσότερες όμως διαμαρτυρίες ε, πέφτουν στο κενό. Πολλές ε, χώρες ε, λένε διάφορα λόγια που δεν εξυπηρετούν καθόλου τους εξεγερμένους. Είχαμε πολλά τέτοια παραδείγματα στη Γουινέα Μπισάο, αλλά δεν αρκούν τα λόγια. Θα πρέπει να αναδείξουμε και να στυλιτεύσουμε την κατάσταση στη Γουινέα Μπισάο, γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, αν δεν γίνει ορατό αυτό το πρόβλημα, θα επαναληφθεί η κατάσταση και στο μέλλον. Και θέλουμε να ε, γίνει προβολή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φτάνουν πια τα λόγια. Είχαμε ένα σχέδιο ψηφίσματος στην ομάδα. Το ίδιο έκαναν και άλλες πολιτικές ομάδες συνέταξαν αντίστοιχα ψηφίσματα, θα πρέπει να πει το λόγο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την κατάσταση που είναι εξαιρετικά σοβαρή. Δεν μπορούμε να μένουμε τα χέρια σταυρωμένα. Αυτή είναι η ώρα για να αναλάβουμε δράση. Και αυτή τη δράση ζητώ και από την είπατε εκπρόσωπο που απουσιάζει στη συζήτηση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς στην ακολουθητή απορία η ακολουθή απορία είναι μια υποστήριξη προς τις νόμιμες αρχές, τις, αρχέ τη αρχές της ε, Γουινέας Μπισά προκειμένου να παταχθεί το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η ανασφάλεια που επικρατεί στην χώρα και στην περιοχή. Αυτό είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και ελπίζω αυτά τα μέτρα να εξαγγελθούν από το Συμβούλιο και από τους ηθήνοντες. Αυτή την πορεία θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Επόμενος αγορητής, είναι ο συνάδελφος κύριος Πίτερ Στασνή για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 12 Απριλίου ο κόσμος έλαβε ανησυχητικές πληροφορίες από την Αφρικανική Ήπειρο. Η στατιωτική οργάνωσαν στη Γουινέα Μπισάου τέσσερα προξικοπήματα για λόγους δίθεν ασφαλείας. Το αποτέλεσμα ήταν βεβαίως το αντίθετο του επιδιωκόμενου στόχου. Η χώρα και η Ήπειρος ε, ε, μαστίζονται από λιγότερη σταθερότητα, φτώχεια και βία. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει, πρέπει να ανατραπεί. Η Γουινέα Μπισάου χρειάζεται εξωτερική βοήθεια. Το Οικονομικό ε, Συμβούλιο, τα Ηνωμένα Έθνη, η Αφρικανική Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Η σταθεροποίηση της χώρας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ένα αποτελεσματικό κράτος δικαίου, βελτίωση της εκπαιδείας και της κοινωνικής συνοχής θα αυξήσουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές. Αν οι στρατιωτικοί της Γουινέας Μπισάο ε, λυπούνται και αγαπούν τους πολίτες τους, πρέπει να ακολουθήσουν το σωστό δρόμο. Αλλιώς η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις και πιέσεις ώστε να τους κάνει να αλλάξουν άποψη. Η δήλωση της κυρίας Άστον της 20 Απριλίου που καταδικάζει στεναρά αυτό το πραξικόπημα είναι ένα από τα πρώτα βήματα προς τη κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ε, δίνω το βήμα τώρα στον συνάδελφο κύριο Φίλιπ Κάτσομαρεκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι το πραξικό, τα πραξικοπήματα κυρίως πλήττουν χώρες με χαμηλά εισοδήματα και ε, βασανίζουν τους πολίτες. Η Γουινέα είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα όπου διεξήχθη πραξικόπημα ε, λίγο πριν το δεύτερο γύρο προεδρικών ε, κλογών πραξικόπημα αντανακλά πολύ αρνητικά και έχει αρνητική επιδράση στους σημαντικότερους ε, τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερα στο εμπόριο Κάσιους, που είναι το 80% των εξαγωγών της Γουινέας Μπισάου. Η συγκομιδή Κάσιους ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου, λίγο μετά το πραξικόπημα, κάτι που έριξε τις τιμές. Οι παραγωγοί λοιπόν προτιμούν να περιμένουν καλύτερες μέρες ε, και δεν θέλουν να πουλήσουν στην αγορά με τόσο χαμηλές τιμές. Μερικοί όσοι τα καταφέρνουν πηγαίνουν στη Σενεγάλη και προσπαθούν εκεί να πουλήσουν τα κάσιους τους. Οι συγκομιδές κάσιους ε, ρυθμίζουν τη ζωή χιλιάδων οικογενειών στο Γουινέμπισαο και απειλούν την ευημερία τους. Δυστυχώς ε, δεν λειτουργεί το κράτο δεν λειτουργούν οι τράπεζε, έχουν ανασταλεί λειτουργία πολλών σημαντικών θεσμών και μάλιστα η προσωρινή ε, άσκηση εξουσίας γίνεται από την αντιπολίτευση με συνεννόηση με το στρατό. Φαίνεται ότι έγινε τέτοια συνεννόηση μεταξύ πραξιοκομματών και αντιπολίτευση. Γι' αυτό και θα είναι πολύ δύσκολη η επαναφορά τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Τελευταίο ομιλητή είναι ο κύριο Ζωάο Φρέιρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και καταδικάζουμε εντόνω το στρατητικό πραξικόπημα στη Γουινέα Μπισάου. Καμία λύση στη χώρα δεν θα είναι αποδεκτή αν δεν αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη και η πολιτική κατάσταση στην Γουινέα Μπισάου χωρίς επεμβάσεις, χωρίς εξωτερικές ε, ε, επιταγές. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα θεσμικά όργανα, τους ε, νόμιμους ε, εκπροσώπους του λαού της Γουινέας Μπισάου και συνέχιση της ε, εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης, θα πρέπει να αποφευθούν οποιασδήποτε αποφάσεις που δεν τηρούν αυτά τα κριτήρια και επιβάλλουν και φέρουν προτελεσμένο γεγονότων την κατάσταση ή παίζουν το παιχνίδι των στρατιωτικών θα πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς πολίτες που έχουν ε, συλληφθεί μετά το πραξικόπημα και θα πρέπει να καταδικάσουμε τα μέτρα που ε, εφαρμόζουν καταστολή ε, ακτιβιστών, πολιτικών ή πολιτών το, της Γουινές Μπισάου που διαμαρτυρήθηκαν για το στρατιωτικό πραξικόπημα. Το πραξικόπημα αυτό και η κατάσταση που επικρατεί έχουν σχέση με κάποια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του λαού της Γουινέα Μπισάου. Θα πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς το λαό αυτό και να απευθύνουμε έκκληση για την ανάληψη κατεπηγόντων μέτρων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του λαού αυτού. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ανησυχητικά μετά το πραξικόπημα στη Γουινέα Μπισάου. Έχουμε καθημερινά απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια. Λείπουν τρόφιμα, δεν υπάρχουν φάρμακα, πόσιμο νερό, ε, καύσιμα. Δεν μπορούμε να γνώμη αυτή την κατάσταση, γιατί ε, πολλοί έχουν ευθύνες ε, για την κατάσταση της χώρας αυτής. Ακόμη και πριν το πραξικόπημα που επιδεινώθηκε με το πραξικόπημα, πέτυχαν τα προγράμματα της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είχαμε τις ε, συμφωνίες υποτιθέμενες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Θέλουμε μια γνήσια συνεργασία που θα απαλύνει τα προβλήματα της χώρας με σεβασμό το δικαίω, του δικαιώματος του λαού να αποφασίσει με κυρίαρχο τρόπο για το πεπρωμένο του. Κασία Κάτς Διάη, έχει σημειωθεί μία μόνο δήλωση βουλήσεως. Η κυρία Έλενα Μπασέσκου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Γουίνεα Μπισάου εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζει ε, με αστάθεια εμπόριων ναρκωτικών ε, και βία. Το πραξικόπημα ανέτρεψε το αποτέλεσμα των εκλογών και επέτεινε, την κατάσταση. Είναι λοιπόν ε, σημαντικό να μην ασκείται πλέον βία ε, να υπάρξει διεθνή συμφωνία για έξοδο από την κρίση και επίσης ε, να μεταβιβαστεί η εξουσία σε ε, πολιτικούς εκπροσώπους. Χρειαζόμαστε μια ουσιαστική πραγματική δημοκρατική μετάβαση. Η αλληλεγγύη της διεθνούς κοινότητας είναι πολύ σημαντική. Εγώ χαιρετίζω ε, το ψήφισμα των εθνών, το 2048 που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα Ηνωμένα Έθνη και ο θετικός ρόλος ε, ε, της Ακοβάς και, αυτή είναι, και αυτός είναι πολύ σημαντικός που καταδίκασε το κρατικό πραξικόπημα. Επίσης απαιτεί την επόμενη εβδομάδα να σταλούν στρατιωτικές δυνάμεις. Ναι, Νικολάη Βάμεν, εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και της Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη για τις ε, πολύ καταρτισμένες παρατηρήσεις τους ε, και για την ανησυχία που εξέφρασαν σχετικά με την κατάσταση στη Γουινέα Μπισάου. Πριν λοιπόν απαντήσω εξ ε, της ε, είπα της εκπροσώπου θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια ε, για το που ακριβώ βρισκόμαστε σήμερα. Ακόμα και η είπατε εκπρόσωπος σε ένα μόνο μέρος μπορεί να βρίσκεται την ίδια στιγμή, όχι σε πολλά. Σήμερα η είπατε εκπρόσωπος βρίσκεται στη Βαγδάτη για να συζητήσει για το πρόβλημα του Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι παρούσα ε, ούτε και ο κύριος Νέσκακ ε, γιατί ε, και αυτός βρίσκεται σε αποστολή στη Μαυριτανία, ο Διευθυντής Αφρικανικών Υποθέσεων. Ομιλώντας λοιπόν για την Γουινέα Μπισάου, αποδείχτηκε ότι τα σχόλιά σας δείχνουν ότι πρέπει να επέλθει το κράτος δικαίου. Οι προτεραιότητες της χώρας πρέπει να είναι η επαναφορά της συνταγματικής τάξης. Να αφαιθούν ελεύθεροι οι κρατούμενοι και να δρομολογηθεί δημοκρατική εκλογική διαδικασία. Το πώς ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά παραμένουν ασαφή. Ε, φοβούμαστε ότι ο συμβασμός ε, δεν επικρατεί ε, Πρέπει να συνεχιστούν λοιπόν οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες έτσι ώστε να επιταχυνθεί η βελτίωση της κατάστασης στη χώρα και αυτό πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, ε, τις πορτογαλόφωνες χώρες και όλους τους διεθνείς εταίρους να διασφαλιστεί ότι η στρατηγική σταθεροποίηση θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κρίσιμα θέματα όπως είναι η εφαρμογή ε, των μεταρρυθμίσεων αγώνα κατά της ατιμορρησίας, των ναρκωτικών ε, και της ε, κοινωνικής ε, ανάπτυξης. Προσβλέπω στο ψήφισμα που θα εκδοθεί από το Κοινοβούλιο για όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος και εμείς ευχαριστούμε κύριε Βάμεν. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση και θα ακολουθήσουν κάποιες ανακοινώσεις. Οι αρμόδιες αρχές της Πολωνίας κατέθεσαν έτοιμα για άρση της ασυλίας του κυρίου Βαλένσα.